Αδελφοί, τότε θα ε, προσθεθεί και αυτή στα πρακτικά της συνεδρίασης. Περνάμε κατόπιν συναρπαστικές ανακοινώσεις του Προέδρου. Σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 6, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών μου είπε πως δεν υπάρχει καμία αντίρρηση έναντι δύο συστάσεων επιτροπών, δηλαδή σύσταση της Επιτροπής ε, Συγκοινωνιών για να μην υπάρξει αντίρρηση σε εφαρμοστικά μέτρα και ακολουθεί βεβαίως και η σύσταση της Επιτροπής Γεωργίας για αναλογαμετρά στον τομέα της Γεωργίας. Οι συστάσεις αυτές θα υιοθετηθούν εκτός εάν κάποια ομάδα ή 40 βουλευτές εντός 48 ωρών φέρουν κάποια αντίρρηση. Εάν όχι ε, θα εγκριθούν εάν ναι, αν υπάρξει αντίρρηση, θα υπάρξει πλειοψηφία. Αν έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βρίσκονται στο Seance undirect. Τον Ιούλιο μετά την διακοπή, όχι, με συγχωρείτε. Τον Ιούλιο μετά την διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7.